Colleagues, good morning. Καλημέρα συνάδελφοι. Να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη σας παρακαλώ πολύ. Την εγκρίναμε. Έγκριση πρακτικών της 20ης και 21ης Ιανουαρίου του 2014. Δεν έχετε αντιρρήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο σημείο. ανακοινώσεις για τις αποφάσεις των συντονιστών της τελευταίας του συνάντησης δηλαδή. Σταθείτε λίγο γιατί δεν έχω το σωστό χαρτί μπροστά μου. Ευχαριστώ λοιπόν απόφαση ότι η ECR θα, έχει, θα μας δώσει τον, τον εισηγητή για γνωμοδότηση της, του προϋπολογισμού. Αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές. Όσον αφορά τους ορισμούς εισηγητών αποφασίστηκε για τον κανονισμό για το άρθρο 120 είπαμε να μην ε, αναλάβουμε ξεχωριστή δράση όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις. Πρόταση για οδηγία για την ε, μείωση κάποιων εκπομπών υπεύθυνη επιτροπή η ΕΝΒΗ. Απόφαση των συντονιστών είναι ότι ε, θα πρέπει η ΕΝΚΟ να αποφασίσει εάν θα έχουμε γνωμοδότηση θα δούμε, θα το δούμε μετά τις εκλογές, αμόλυνση των οχημάτων. Έχουμε την έκθεση, την ενδιάμεση έκθεση για το, τα ομόλογα έργου 2020. Ε, καλούμε την Επιτροπή, θα καλέσουμε μάλλον την Επιτροπή να κάνει μια παρουσίαση για το θέμα αυτό σε κάποια επόμενη συνεδρίαση. άλλες ε, εκθέσεις, ε, γαλάζια ενέργεια, δραστηριότητες ε, γενική έκθεση της ΑΦΚΟ. Επίσης, ε, ε, το, κλίμα, το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς επίσης και μείωση μολυντικών εκπομπών, θα αποφασίσει η Επιτροπή από αυτού αργότερα. Επίσης, ε, οι συντονιστές έλαβαν γνώση της επιστολής επιτροπολογίας 4-5 μετά από μακρά συζήτηση αποφάσισαν οι συντονιστές να δεχτούν ε, την προσέγγιση που προτείνει η επιστολή Κάλλας στα διάφορα οι συντονιστές αποφάσισαν να ε, μην ε, γίνει μέχρι την επόμενη συνεδρίαση ε, η αποτίμηση των, μεγάλων, των επιπτώσεων των μεγάλων πλοίων, των Giga Liners. Τίποτα άλλο. Ερωτήσεις όσον αφορά τους συντονιστές. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλά ήθελα να σημειώσουμε ότι στη συνάντηση των συντονιστών για την λήψη απόφασης σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις του κανονισμού Connecting Europe, διασυνδέοντας την Ευρώπη. Είναι θέματα που χαίρομαι που ελήφθη αυτή η απόφαση και την θεωρώ σωστή και βαίνει καλός και θα ήθελα να υπήρχε πρόσκληση για συμμετοχή σε αυτή τη συνεδρίαση. Να μην νομίζει η Επιτροπή ότι όταν παρίσταμε υπάρχουν προβλήματα και όταν απουσιάζω δεν υπάρχουν προβλήματα, διότι διαφορετικά δεν θα είναι καλό αυτό για την ε, ε, κατάσταση γενικότερα. Αλλά για την ε, υποστήριξη από την Επιτροπή θα προτιμούσα να ήμουν παρούσα κατά, την, κατά τη στιγμή η λήψη απόφαση υπέρ και είμαι υπέρ. Απλά να σημειώσω ότι υπάρχει ένα σημαντικό σφάλμα στα ισπανικά στο ε, κεφάλαιο 6 στο άρθρο 17 όπου λέγεται ότι τα, πολι... τα πολιετή προγράμματα θα υιοθετηθούν μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων. Δεν γίνεται έτσι, αλλά μέσω εκτελεστικών πράξεων. Απλά και μόνο να σημειωθεί αυτή η ανάγκη, να τροποποιηθεί δηλαδή αυτό στη διατύπωση στα ισπανικά, στο κεφάλαιο 6, στο αεδάφιο, ε, στο άρθρο 17. Ευχαριστώ. Θα το δούμε αυτό. Θα δούμε λοιπόν και ούτως ή άλλως ε, δεν ε, ήθιστε, ε, εν πάση περιπτώσει, συνήθως οι Γερμανοί κάνουν προβλήματα, αλλά πάντως το σημειώνουμε αυτό που είπατε. Τίποτα άλλο, όχι, επόμενο σημείο επομένως είναι... My notes. German's notes now for the meeting. Είναι η ψηφοφορία. So, this is the Ναϊάδες 2 λοιπόν. Η συγητή, μάλλον η συγήτρια η κυρία Βόρτμαν Κόλ, Ξεκινάμε κάνοντας έναν πρώτο έλεγχο, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Τρέξε, τρέξε, προλαβαίνεις. all the right read the titles what we are voting so that they know because we have a few small... Vote closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Είμαστε όλοι εντάξει. Επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρόταση κανονισμού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό 718 του 1999 σχετικά με την μεταφορική ικανότητα των κοινοτικών στόλων στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Μου είπαν ότι πρέπει να διαβάσω τον τίτλο της έκθεσης. Στις πρώτες τρεις τροπολογίες δεν έχουμε να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αποσχόληση 5 υπέρ κατά αποχέσε Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας τη ψηφοφορία. Και απερίφθη. Απασχόληση 6. Υπέρ. Κατά. αποχέσε Απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. Συμβιβασμός 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 8. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά προτιμώ να ελέγξουμε. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Και απερίφθη. Τελική ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 30 ε, υπέρ, μία ψήφος κατά, δύο αποχές, νομοθετικό ψήφισμα υπέρ. Ε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Το ίδιο αποτέλεσμα, 30 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, δύο αποχές, επομένως εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα ε, την απόφαση για διαθεσμικές διοργανικές ε, συμφωνίες. Θέλετε ηλεκτρονικά. Εντάξει. Οκ, η ηλεκτρονική ψηφοφορία ξεκινάει. Δεν εμπιστεύεστε την κρίση μου φαίνεται και τα μάτια μου. 32 υπέρ, μία, ε, μία ψήφος ε, ε, κατά καμία αποχή και με τη βούλα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας λοιπόν. Προχωράμε. Δέκτερη έκθεση της Κορίν Cool πρόταση οδηγίας ε, για τις τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοείας που καταργεί την οδηγία 2006-87-ΕΚ ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τροπολογία 16, άρθρο 5, παράγραφος 2 της κυρίας Τικάου υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 1 του κυρίου Φιντάντσα υπάρχει κάποιος που αντιτίθεται όχι άρα ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 είναι γλωσσική, τροπολογία 9 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία της κυρίας Τικάου. Αντιτίθεται κάποιος στην προφορική αυτή τροπολογία. Όχι, επομένως την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 19 κατά, καμία αποχή, 14 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ε, σαν προσθήκη στο κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 3 της εισηγητρίας ε, δεν φαίνεται να διαφωνείτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 32 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λείπουν μερικέ ψήφοι. Τώρα εντάξει, πέρασε τι προφορίε, 31 ψήφοι υπέρ, μία ψήφο κατά καμία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Βόρτμαν Κόλ. Περνάμε τώρα στην απαλλαγή 2012 Γενικός Προϋπολογισμός τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι κάνουμε, αλλάζουμε οδηγούς, συνοδηγούς εδώ. Ωραία. όχι, όχι, μένουμε με την ίδια ομάδα. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η μία καταπίπτει, συμβιβασμός 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 της κυρίας Ντουιρόν, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία από τον εισηγητή έχετε καμία αντίρρηση όχι άρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επί της παραγράφου 9 έχουμε μια χωριστή ψηφοφορία, η πρώτη μέχρι από Proposed That Year 2012, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, as soon as μέχρι κορτοβόντιτος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 4 κατά καμία αποχή, επομένως εγκρίνεται. Επόμενη απαλλαγή 2012 σχετικά με την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Πάντα για το 2012 εισηγητής ο κύριος Νταντάν, τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, κατά τμήματα ψηφοφορία που έχει ζητηθεί από, τους, ε, την Άλντε, μέχρι single seat, υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είμαι σίγουρος, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πρώτο τμήμα λοιπόν. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 25 ψήφοι υπέρ 4 κατά 3 αποχές. Δεύτερο τμήμα, το υπόλοιπο του κειμένου. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει πάρα πολύ λογική, γιατί στο πρώτο τμήμα ζητήσαμε ε, μία έδρα και στο άλλο μία τοποθεσία. Εν πάση περιπτώσει, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Οι 26 ψήφοι υπέρ 4 κατά καμία αποχή επομένως εγκρίνεται. Επόμενο πάλι του κυρίου Νταντάν, σχέδιο γνωμοδότηση για την απαλλαγή του Σέζαρ. Μία τροπολογία μόνο, της κυρία Τικάου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 30 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή, επομένως εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην απαλλαγή όσον αφορά την υλοποίηση του ε, προϋπολογισμού της ΕΜΣΑ υπέρ του τροπολογίας 1. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ. Κατά Αποχέσε, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 29 ψήφοι υπέρ 3 κατά καμία αποχή, επομένως εγκρίνεται και φτάνουμε πάλι στην ε, γνωμοδότηση του κυρίου Νταντά σχετικά με την απαλλαγή ε, για το έτος 2012, ε, υλοποίηση του, κανον, του προϋπολογισμού για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι της ψηφοφορίας 28 ψήφοι υπέρ 4 ψήφι κατά καμία αποχή επομένως εγκρίνεται μπράβο και έβγε σας κύριε Μισελ Ντόντα να πω ότι ο κύριος ε, ε, Κουσιέρη γίνεται, ε, έχει γενέθλια σήμερα. Συγχαρητήρια. So next is the presentation of the 2014 draft Λοιπόν, θα έχουμε τώρα παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα προγράμματα εργασίας ΔΕΔΕΜ για το 2014 από τη Γενική Διεύθυνση MOVE. Ε, βεβαίως μπορούν να μείνουν όλα τα μέλη, αλλά επειδή είναι και κλεισμένο το...